έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι προσπάθεια ε, γίνεται για να ε, ζήσει ο λαός της περιοχής εν ειρήνη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κλείνουμε τώρα τη συζήτηση. Έξι προτάσεις ψηφίσματος έχουν κατατεθεί, θα ψηφιστούν στις 12 την Πέμπτη. Προχωρούμε τώρα στην εξέταση της έκθεσης Κοέλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου Σέγγεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Καλωσορίζω την Επίτροπο και δίνω το λόγο στον κύριο Κοέλιο ως εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, συνάδελφοι, κάποιες παρατηρήσεις πρώτον. Ενίσχυση του Σέγγεν. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων είναι μια, μια από τις βασικές επιτυχίες και επιτεύγματα της Ένωσης και ένα βασικός πυλώνας της Ένωσης. Για το λόγο αυτό θεωρούμε, όπως και άλλοι, ότι δεν πρέπει να αποδυναμωθεί. Αντίθετα, πρέπει το Σέγγεν να ενισχυθεί και να προστατευτεί. Αυτή τη θέση πήρε και η κυρία Μάλιστο, μάλιστα πριν από λίγο και Ξεκινήσαμε με πέντε κράτη, πέντε ιδρυτικά κράτη της Ένωσης στο Σέγγεν και ακολουθήθηκε, ωστόσο προσχώρησαν σιγά σιγά ε, άλλα 25 κράτη της Ένωσης και όχι με, 700, με, ε, με 7.000 ε, ε, χιλιόμετρα χερσαία σύνορα. Δεύτερη παρατήρηση. Αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η κατάργηση των εσωτερικών σύνορων απαιτεί αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του SIS, καλή αστυνομική συνεργασία και ανάγκη αποτελεσματικών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα. Η ασφάλεια του χώρου Σέγγεν εξαρτάται από την αυστηρότητα και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα από κάθε κράτο. Όταν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αποδυναμώνεται ολόκληρο ο χώρο Σέγγεν, υπονομεύεται η αξιοπιστία τη Ένωση και καταστρατηγείται η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τρίτη παρατήρηση. Η ισότητα κανόνων για όλους. Η εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρχει και στις διαδικασίε που θα πρέπει να είναι σαφείς και δίκαιες. Οι υποψήφιε χώρε θα πρέπει να εφαρμόζουν με αποτελεσματικό και σωστό τρόπο όλα τα κριτήρια του Σέγγεν. Τα ίδια κριτήρια που χρειάστηκε να τηρήσουν κατά ανάγκη και οι προηγούμενε υποψήφιε χώρε. Ούτε περισσότερου κανόνε ούτε λιγότερου. Τέταρτον, διαφάνεια στο όνομα της ελευθερίας αλλά και στο όνομα της ασφάλειας θα πρέπει να παρέχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Με λυπή που εκ νέου το Συμβούλιο δεν συμπεριφέρθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανούμενο την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις εκθέσεις αξιολόγησης. Το πρόβλημα θα μπόρεσε να ξεπεραστεί μόλις, ε, μόνο χάρη στον ζήλο των πρέσβεων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας που ζήτησαν να πάψουν οι εκθέσεις να έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και να αποσταλούν στο Κοινοβούλιο, επιτρέποντας έτσι τα μέλη του Κοινοβουλίου να έχουν πρόσβαση στην αξιολόγηση των συστάσεων. Το Συμβούλιο εκ νέου δεν έδειξε σεβασμό προς το Κοινοβούλιο. Η ίδια διαφάνεια απαιτείται και λόγω των κρεμών προβλημάτων που αναφέρθηκαν, που μπορεί να μην αποτελούν εμπόδιο για την πλήρη ένταξη στο Σέγγεν των δύο αυτών χωρών πρέπει ωστόσο να αποτελέσουν αντικείμενο μιας συνοδευτικής προσέγγισης και μιας βοήθειας από την Επιτροπή αξιολόγηση. Πέμπτο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Είπαμε τόσες φορές για την αξία της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Από τη στιγμή της ένταξής τους στην Ένωση το 2007, η Ρουμανία και η Βουλγαρία ήλπιζαν θεμητά να γίνουν οι πολίτες, τους Ευρωπαίοι πολίτες και να απολάβουν έτσι όλων των δικαιωμάτων που απολάβουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, κυρίως στην ελευθερία κυκλοφορία στο πλαίσιο του χώρου Σέγγεν. Και έκαναν καλή δουλειά. Και οι δύο χώρες αξίζουν συγχαρητήρια από πλευρά μα για όλα όσα πέτυχαν, αλλά και δέσμευση που ανέλαβαν να υλοποιήσουν στο μέλλον για να μπουν στο Σέγγεν. Αυτό προκύπτει και από τις εκθέσει αξιολόγηση και από, την αποστολή, και από τις αποστολές της δύο χώρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκου και Έντσιου αλλά και του, του, του συναδέλφου ε, Κόβατσο και Νεντέλτσεβ από τη Βουλγαρία για τις συνεργασίες τους. Με χαρά θα δεχθούμε τις δύο χώρες των χώρο Σέγγεν και ελπίζω ότι το Συμβούλιο όταν λάβει την τη θέση μας να ακολουθήσει την ίδια θέση. Τον λόγο τώρα εξ του Συμβουλίου έχει η κυρία Γκιόρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητά μέλη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα να συμμετέχω στη διεύρυνση της ζώνης Σέγγεν προς Βουλγαρία και Ρουμανία. Αυτή ήταν μια βασική προτεραιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας. Ε, βλέπω με ευχαρίστηση ότι και η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν λάβει θετικές εισηγήσεις από τις τεχνικές ομάδες σχετικά με την εφαρμογή του συνόλου του κεκτημένου Σέγγεν και η δική σας φυσικά εξέταση του θέματος έχει οδηγήσει στα ίδια αποτελέσματα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Καύλος Κοέλιο για την επαγγελματική αρτιότητα της προσπάθειάς του. Να θυμίσω εδώ ότι όταν η Ουγγαρία από την Κεντρική Ευρώπη ενετάχθησαν στο Σέγγεν ε, υπήρξε μια τεχνική δυσκολία σχετικά με την ανάπτυξη του CIST, του τεχνικού συστήματος. Και τότε η Πορτογαλική Προεδρία ήταν αυτή η οποία είχε εφεύρει, θα έλεγε κανείς, τη λύση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τον πρόεδρο της Αρμόδιας Επιτροπής, της Επιτροπής Λίμπε, τον κύριο Λόπε Αγουιλάρ, για την προσπάθειά του. Η Ουγγρική Προεδρία έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για να προχωρήσει η διαδικασία. Η Προεδρία είπε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν κάποιες αμφιβολίες και επιφυλάξεις από πλευράς των κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε προσπάθεια. Το θέσαμε στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης του Συμβουλίου Τζάι στις 23 και 24 Φεβρουαρίου και εκεί το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα της Προεδρίας για την ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας σε στενή συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη για να καταλήξουμε σε μια λύση των προβλημάτων αποδεκτή από όλους. Αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία και η Ρουμανία πήραν τα απαιτούμενα βήματα έτσι ώστε οι πολιτικές και οι πρακτικές τους να είναι συμβατές με τα επίπεδα του Σέγγεν και περιλαμβάνονται εδώ τομείς όπως προστασία δεδομένων, αστυνομική συνεργασία, έλεγχος εξωτερικών συνόρων, έκδοση θεωρήσεων και αποτελεσματική εφαρμογή του CIS. Ταυτόχρονα, η αφομοίωση των Σέγγεν, από, μάλλον του Σέγγεν σε επίπεδο όλων των κεφαλαίων από, τις χώρες, από τις δύο χώρες ε, κατέληξε θετικά. Πήραμε το OK και από την τεχνική ομάδα και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή στα πλαίσια του Τζάι, του Συμβουλίου Τζάι. Γνωρίζω ότι κάτι τέτοιο ε, είναι ιδιαίτερα επιθυμητό για πολλούς από εσά. Και για, ιδίως για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη συμμετοχή τους στο Σέγγεν. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο σε όλους τους τομείς καθότι η σωστή συνέχεια αποτελεί μια μόνιμη διαδικασία σε όλες τις χώρες Σέγγεν. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω στο πλαίσιο αυτό ότι και η Βουλγαρία και η, Βουλγαρία, και η Ρουμανία θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν τακτικές εκθέσεις για τα βήματα που έχουν λάβει για να αντιμετωπίσουν προβλήματα, τυχόν προβλήματα. Ιδίως στην, ε, στους ελέγχους στα σύνορα και την, και την αστυνομική, διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία καθώς και το θέμα της έκθεσης, της έκδοσης θεωρήσεων. Όταν εγκρίνεται στην την έκθεση Κοέλιο και το Συμβούλιο υιοθετήσει τα συμπεράσματα της Προεδρίας, το μόνο που θα μένει είναι η ομοφωνία στο Συμβούλιο. Το υπογραμμίζω ότι το Συμβούλιο μπορεί να επανέλθει σύντομα στο θέμα για να εξετάσει πώς μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία ίσως το Σεπτέμβριο φέτος. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κύριου Κοέλιο θίγει το ζήτημα της πρόσβασης στα εμπιστευτικά έγγραφα. Το ανέφερε και στα σχόλιά του εισηγητής. Ένα σημαντικό θέμα όταν εξετάζαμε το ζήτημα. Η πρόσβαση του Κοινοβουλίου στα εμπιστευτικά ε, ε, έγγραφα είναι από τα εκκρεμή διοργανικά θέματα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου που προτίθεται να επιλύσει η Προεδρία, η Ουγγρική Προεδρία. Προχωρήσαμε, βρήκαμε το δρόμο με την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, ωστόσο η γενική λύση του θέματος θα πάρει χρόνο. Η Προεδρία από το ξεκίνημά της προσέβλεπε σε μια άμεση λύση του ζητήματος για να μην υπάρχει καθυστέρηση της πρόσβασης των δύο χωρών στο χώρο Σέγγεν. Στο ίδιο πλαίσιο, κατόπιν προτάσεως της Ουγγρικής Προεδρίας, το Συμβούλιο έδωσε την συγκατάθεσή του, τόσο ώστε το Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση στα κείμενα που σχετίζονται με την προσχώρηση των δύο κρατών μελών στην ζώνη Σέγγεν. Συνολικά, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η, Προεδρία, η Ουγγρική Προεδρία είναι πεπισμένη ότι η διεύρυνση του χώρου Σέγγεν με τι δύο χώρε, τώρα που πληρούν τους, τα τεχνικά και νομικά κριτήρια, θα είναι θετικό για όλη την συνεργασία της ζώνης Σέγγεν και για την Ευρώπη. Α, για μια ελεύθερη Ευρώπη από την Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον Ατλαντικό χωρίς να δείχνει κανείς διαβατήρια και μην ξεχνάτε ότι όντως η ελευθερία κυκλοφορίας είναι ένα από τα βασικά θεμέλια της Ένωσης, απτό για τον πολίτη και κάτι που όλοι επιζητούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Επιτροπής, η κυρία Μάλμσον. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Το Σέγγεν είναι ένα καταφληκτικό επίτευγμα. Είναι τα πιο απτά ε, δώρα που δίνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στου πολίτε, όπω είπε ο ε, εκπρόσωπος Προεδρία, μπορεί να πάει κανένα από τη Φιλανδία στην Πορτογαλία χωρί να σταματά σε ελέγχου στα σύνορα. Ε, θα πρέπει να σταματήσουν οποιασδήποτε προσπάθειε για επανεισαγωγή δώρο. και πολλέ φορέ συζητήσαμε πώ θα μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε το Σέγγεν και όχι να το αποδυναμώσουμε. Θέλουμε περισσότερο Ευρώπη και λιγότερη Ευρώπη. Θα καλύτερη αξιολόγηση, καλύτερα μέσα για καλύτερες κατευθύνες γραμμές και συστάσεις πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί το κεκτημένο Σέγγεν. Και αυτό συζητηθεί αυτή την εβδομάδα με τα κράτη-μέρη στο Συμβουλίο. Αλλά και στην ε, διάσκεψη κορυφή τέλη Ιουνίου. Δεν θέλω να συγχαρώ την Βουλγαρία και την Ρουμανία για τις προσπάθειες που κατέβαλαν. Τα είδα εγώ ήδη η ότι κατέβαλαν σημαντικότητε ε, προσπάθειες και είχαν το πλεονέκτημα να εκμεταλλευτούν τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και με εντυπωσίωση ο τρόπος με τον οποίο το έκαναν. Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ την ε, Ρουμανία και την Βουλγαρία για τις προσπάθειες αυτές. Το αποτέλεσμα είναι ότι και οι δύο μπορούν να πληρούν τα τεχνικά κριτήρια του Σέγγεν και κατέδειξαν ότι είναι πραγματικά θεσμευμένοι για να αξίζουν την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν χαιρετίζει λοιπόν αυτή την έκθεση και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όχι μόνο τις δύο χώρες αλλά και τον κύριο Κοέλιο και τους κοιόδους ηγητής για την έκθεση αυτή. Πάντα η Κομισιόν θεωρούσε ότι δεν υπάρχει επίσημο σχετισμό μεταξύ του μηχανισμού CBM και του συμφωνία Schengen, τη έναξη του Schengen. Όλοι ξέρουμε όμω ότι αυτή η πρόσβαση βασίζεται σε εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη, η έλλειψη εμπιστοσύνη ήταν κάτι που συζητήθηκε πολύ στι περισμένε εβδομάδε η απόφαση να έρθουν τα ιστορικά σύνορα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία θα πρέπει να βοηθήσουν όχι μόνο στην τεχνολογική αξιολόγηση αλλά και στην εμπιστοσύνη αυτή που δυστυχώ δεν υπάρχει σήμερα. Γι' αυτό, όπω είπε και η Προεδρία, θα πρέπει να εργαστούμε στενά με τα κράτη-μέλη για να βρεθεί μια γλίγορη και καλή λύση. Αυτό θα πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητα το Συμβούλιο που είναι εκείνο που αποφασίζει επί του θα πρέπει να ορίσει ένα σαφές πλαίσιο με σαφές προθεσμίες ούτω ώστε η Ρουμανία και η Βουλγαρία να μπορέσουν να προχωρήσουν προς το εμπρός. Απέδειξαν ότι είναι έτοιμες να συνταχθούν, ότι έκαναν τις απαραίτητες προσπάθειες, πέτυχαν τα απαραίτητα και θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να προχωρήσουν και στο Συμβούλιο προ την κατεύθυνση τη απόφαση αυτή Ευχαριστώ. Των ομάδων, ο Δεμέρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον κύριο Κοέλιο και να τον συγχαρώ διότι πραγματικά πάντα ήταν λιτό. Να προσθέσω, πρέπει να βοηθήσουμε τι δύο χώρε. Έχω εμπιστοσύνη στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Δούλεψαν καλά και πρέπει να λάβουν αυτό που δίκαια τους αντιστοιχεί. Δεν είναι δώρο. Το είπε η Προεδρία του Συμβουλίου, αλλά και η Επιτροπή, κύριε Μάρτσον, τηρούν από τεχνικής και νομικής απόψεως τις προϋποθέσεις. Και εγώ συμφωνώ μαζί τους. Δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη άλλα κριτήρια που δεν είναι αυτά που είναι αποκλειστικά τεχνικά ή νομικά. Τα κριτήρια αυτά είναι πέντε Πρώτον, τηρούν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων, τηρούν το σύστημα πληροφόρησης έγκεν, τηρούν την αστυνομική συνεργασία, τηρούν την έκδοση θεωρήσεων και τηρούν τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, είτε είναι χερσαία, είτε θαλάσσια, είτε εναέρια. Επίσης, τηρούν το SIS και το SIREN. Για, όλο, για όλους αυτούς τους λόγους, το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει ένα ανεπιφύλακτο μήνυμα προς το Συμβούλιο, ιδίως δε προς τις μόνιμες αντιπροσωπείες πέντε χωρών που δεν τις αναφέρω τώρα, που τους ξέρουμε, τις ξέρουμε όλοι όμως. Κυρίες και κύριοι, η συμπερίληψη στο χώρο Σέγγεν που έχει πάνω από 400 εκατομμύρια άτομα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας δίνει συν, δεν δίνει πλην. Φτιάχνουμε περισσότερη Ευρώπη. Δεν πρέπει να έχουμε διπλά επίπεδα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να ζητούμε από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να τηρούν όρους που δεν απαιτήσαμε από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη για να είναι στον χώρο αυτό ελευθερίας. Άρα, κλείνοντας, επιθυμώ ανεπιφύλακτα να περάσει ένα ισχυρό πλειοψηφικό μήνυμα από το Κοινοβούλιο προς το Συμβούλιο. Αυτά ευχαριστώ και συγχαρητήρια εκ νέου προς τον κύριο Κοέλιο αλλά και την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κοέλιο για την προσπάθειά του και την εμπειρογνωμοσύνη που προσέφερα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Ουγγρική Προεδρία και την Επίτροπο κυρία Μέλστρομ για την υποστήριξή της. Η συζήτηση για την διεύρυνση των Σέγγεν προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι μια συζήτηση η οποία είναι κυρίως πολιτική και ίσως κάποιοι να ξέχασαν το τι πραγματικά συζητάμε. Στην ουσία εμείς διευκρινίζουμε ε, ότι κάποιες χώρες θα πρέπει να εκπληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για να ενταχθούν στο Σέγγεν. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα δεοντολογικά ή νομικά τα οποία να επιτρέπουν οι κανόνες να αλλάξουν. Οι κανόνες θα πρέπει να βελτιωθούν ίσως μέσω της δημιουργίας του νέου μηχανισμού αξιολόγησης του Σέγγεν που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες και δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να αναγνωρίσουμε ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για ότι δεν πηγαίνει καλά σε ορισμένες χώρες γύρω από τις υποθέσεις αυτές. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν φταίει η Ρουμανία και η Βουλγαρία που είναι υπεύθυνε για το ότι ορισμένες χώρες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τα σύνορά τους και τις μεταναστευτικές ροές. Δεν είναι υπεύθυνη η Ρουμανία και η Βουλγαρία για τις τάσεις που ακολουθούν ορισμένες κυβερνήσεις οι οποίες θέλουν να εφαρμόσουν αντιμετασταυτικές πολιτικές ιδιαίτερα εις βάρος των ε, πολιτών Ρωμά. Και τέλος, οι πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας δεν θα πρέπει να ε, υποφέρουν λόγω των κακών σχέσεων που έχουν ε, κάποιες ε, χώρες ή κάποιοι ηγέτες μεταξύ τους. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να σεβαστούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λειτουργήσει αυστηρά ως θεματοφύλακα συνθήκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, μιλάμε για ένα θέμα το οποίο φέρνει στην επιφάνεια και πρακτικά προβλήματα αλλά και θέματα αρχής. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο, τον εισηγητή, για τον επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το θέμα αυτό στα πλαίσια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ οι βασικές κοινοτικές αρχές έγιναν δεκτές, έγιναν σεβαστές. Χαίρομαι λοιπόν για το επικοδομητικό πνεύμα του κυρίου Κοέλιο. Έχουμε εδώ λοιπόν ένα θέμα αρχής όταν λέμε πως όταν δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπληρώσουν τα κριτήρια να γίνουν μέλη του Σέγγεν τίθεται το ερώτημα αν θα γίνουν μέλη του Σέγγεν ή όχι. Μα προφανώς ο κανόνας λέει ναι ότι και οι δύο χώρες αξιολογήθηκαν σε σχέση με το επίπεδο προπαρασκευής τους και τα συμπεράσματα είναι κατηγορηματικά θετικά. Ο εισηγητής έκανε ένα βήμα προς τα εμπρός ένα βήμα επιπλέον, πήγε στην, Ισπαν... στην Ρουμανία και την Βουλγαρία συνοδευόμενος από, τον... από τους συνεισήγητές τους για να δει πώς εξελίσσονται τα θέματα στα εξωτερικά σύνορα σαν παράδειγμα. Υπάρχει επίσης το θέμα των θεσμικών σχέσεων ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι κάποιοι ε, ευρωβουλευτές θα έπρεπε να έχουν την πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα εμπιστευτικά, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Αυτό έγινε αντικείμενο σκληρής κριτικής από πλευράς της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και ε, ε, χαίρομαι γιατί πράγματι επικράτησαν απόψεις και αντιλήψεις οι οποίες είναι σωστές. Οι απαιτήσει λοιπόν των θεσμικών οργάνων και των χωρών θα πρέπει να είναι δημοκρατικές και έλογες. Νομίζω ότι η ψηφοφορία γύρω από το θέμα αυτό θα, θα δώσει το πράσινο φως στην ένταξη των δύο αυτών χωρών στο χώρο Σέγγεν. Uh, ε, κύριε Επίτροπε, Κύριε οι Ευρωπαίοι πολίτες χάνουν όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη τους απέναντι στα κοινοτικά προγράμματα. Δεν θα πρέπει να το παρατραβήξουμε εφόσον δεν είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Αυτό το αίσθημα έχουν πολλές χώρες όσο ό,τι αφορά το χώρο Σέγγεν. Να μην ε, σπεύσουμε να διευρύνουμε περαιτέρω το χώρο, δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Βέβαια, δεν θα πρέπει η συζήτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ω ε, άλοθη, ω πρόσχημα να επικρίνουμε τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, γιατί πάσχησαν για να εκπληρώσουν τα τεχνικά κριτήρια που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να διαφωνούμε βέβαια ω προ το κατά πόσο εκπληρώθηκαν τα κριτήρια αυτά. Σίγουρα έγινε μεγάλη πρόοδο από τι δύο χώρε. Πάντω είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για την ανανέωση τη εμπιστοσύνη του συστήματο Σέγγεν και την ακαιρεότητα τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ευκαιρία να να ολοκληρώσουμε έναν ενημερωμένο και αποτελεσματικό μηχανισμό αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε τι τρέχουσε ούτε τι μελλοντικέ προκλήσεις ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να θεσπίσουμε κάποια κριτήρια που δεν θα καλύπτουν μόνο τα τεχνικά στοιχεία του συστήματος έγκαινα, αλλά θα αξιολογούν τον αντίκτυπο του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, ε, ακόμη και στις αξιολογήσεις των μελών της, του χώρου Σέγγεν. Θα πρέπει να προβούμε σε νέες αξιολογήσεις και ένας νέος μηχανισμός ίσως θα γεφυρώσει την έλλειψη εμπιστοσύνη που υπάρχει αυτή τη στιγμή που ακούμε ε, όχι μόνο εντός του Μικυκλίου αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. President, Honorable Commissioner... Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα είναι αν θα εγκρίνουμε την προσχώρηση στο χώρο Σέγγεν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Και εγώ κατάγομαι από νέα χώρα μέλος και θυμάμαι πόσο επιθυμούσαμε διακαώς να μπούμε στο χώρο Σέγγεν. Γι' αυτό και με υπέρ τη ένταξη στο χώρο Σέγγεν τη Ρουμανία και τη Βουλγαρίας. Υπάρχουν βέβαια κάποιε αδυναμίε, υπήρξαν κάποια προσκόμματα, αλλά έχουν υπερκεραστεί και οι δύο χώρε είναι πανέτοιμε να προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν το 2011. Αντιλαμβάνομαι τι επιφυλάξει προ τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Γι' αυτό όμω ακριβώ η συνεργασία στα πλαίσια του μηχανισμού συνεργασία και εξακρίβωση θα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε όμως να επινοήσουμε νέα κριτήρια για την προσχώρηση στο χώρο Σέγγεν. Δεν μπορούμε να υπονομεύουμε τη βεβαιότητα ότι μία χώρα θα προσχωρεί εφόσον πληρεί τα υφιστάμενα κριτήρια. Η συζήτηση στο Κοινοβούλιο έδειξε την επιτακτική ανάγκη της αποφυγή διπλών μέτρων και σταθμών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν, σε ό,τι αφορά και τα υπάρχοντα κράτη-μέλη και τα μελλοντικά. Είναι σημαντικό το θέμα της αξιολόγησης. Είναι παράδεκτο ότι ορισμένες χώρες μέλη στο Συμβούλιο πρότειναν την τροποποίηση της νομικής βάσης της πρότασης αυτής, ώστε να αποκλειστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη διαδικασία, διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πάντως ευελπιστώ ότι ο εισηγητής μας, ο κύριος Κοέλιο, θα προασπίσει τα προνόμια και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως κάνει άλλωστε με την αμέριστη υποστήριξή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο για το έργο του και επαναλαμβάνω προσβλέπουμε σε περαιτέρω ε, αγαστή συνεργασία και στο μέλλον. Για και κύριοι, ε, νομίζω έχει φτάσει πλέον η στιγμή η Βουλγαρία και η Ρουμανία να συμπεριληφθούν στην πλήρη εφαρμογή του, ε, της Συμφωνίας Σέγγεν. Η κατάργηση των ιστορικών συνόρων και η ελεύθερη μετακίνηση είναι από τα σημαντικότερα επιτεύγματα και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω πως ορισμένα κράτη μπλοκάρουν αυτή την εξέλιξη, μεταξύ αυτών βέβαια και η Γερμανία. Και προβάλλουν το επιχείρημα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ε, δωροδοκία. Πολλοί λένε ότι θα υπάρξουν ε, ανεξέλεγκτες ροές ε, μετανάστευσης. Εγώ δεν τα κατανοώ αυτά. Αυτό το παιχνίδι που γίνεται με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι πολύ επικίνδυνο. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο εμείς ευθύ εξ αρχή στηρίξαμε τον εισηγητή τον κύριο Κοέλιο και είπαμε ότι για όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπάρχουν οι ίδιες προδιαγραφές και όσον αφορά την εφαρμογή της συνθήκης του ε, Σέγγεν. Και όπως και όλοι οι άλλοι ε, συνάδελφοι στην Επιτροπή μας, εκπλαγήκαμε τα μάλα από τον τρόπο με τον οποίο μας ε, συμπεριφέρθηκε το Συμβούλιο, το οποίο μάλιστα αρνήθηκε να μας διαθέσει τα απαραίτητα έγγραφα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Εμείς θέλουμε η Συμφωνία Σέγγεν να εφαρμοστεί αμελητή και να μην περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Ε, θα ήθελα να παραθέσω την κυρία Φάτη, γνωστή δημοσιογράφος. Οι Ρουμάνοι είναι αισιόδοξοι πολίτες, ε, έχουν στρέψει το βλέμμα στην Ευρώπη και θέλουν να φτάσουν στο επίπεδο των υπόλοιπων κρατών. Εάν λοιπόν τους στρέψουμε την πλάτη, πολλοί ε, θα γίνουν ευρωφοβικοί. Αυτά ισχύουν για την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το άρθρο 4, η παράγραφος 2 της ε, Συμφωνίας Προσχώρησης στο Σέγγεν προβλέπει ότι οι διαδικασίες ελέγχου ε, για, την, για το κατά πόσον εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ε, για την εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφασίσει το Συμβούλιο να καταργήσει τα εσωτερικά σύνορα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να ισχύουν αυτές οι προδιαγραφές. Ε, οι διαδικασίες είναι διαδικαστικής φύσεως και οι διαδικασίες αυτές θεωρούν ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία μπορούν να θέσουν εν κινδύνο την ασφάλεια των υπολείπων κρατών. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις ε, ε, στην ε, θάλασσα, στον αέρα, στην ξηρά όσον αφορά τους ελέγχους και οι αστυνομικέ αρχές δεν μπορούν να ελέγξουν τους παράνομους μετανάστες που έρχονται από αυτές τις δύο χώρες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω να ανασταλεί η διαδικασία ένταξη της Βουλγαρίας και τη Ρουμανίας στη Συμφωνία Σέγγεν με βάση την αρχή της πρόληψης Σκείται βέβαια τεράστια πίεση ε, στα εξωτερικά σύνορα αυτών των ε, χωρών ε, γιατί οι χώρες αυτές τελικά μπορεί να γίνουν παράνομες εισοδοί παράνομων πάλι μεταναστών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, στο ψητό αμέσως. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ως διεφθαρμένα ανατολικά κράτη δεν αξίζουν καθόλου να μπουν στο Σέγγεν. Επαναλαμβάνω, δεν αξίζουν καθόλου. Ωραία τα ιδεαλιστικά που μας λένε οι επίτροποι για το Σέγγεν και παρά τη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου που θεωρεί ότι θα είναι καταπληκτικό να μπουν ε, στο Σέγγεν η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι πεδαριώδες και αφελέστατο. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν δείξει περίτρανα ότι δεν αξίζουν να μπουν στο Σέγγεν. Σύμφωνα με τη διεθνή διαφάνεια και στις δύο χώρες ακόμα είναι καθημερινή υπόθεση ε, ε, η διαφθορά. 3,6 ε, στα 10 και 3, η Βουλγαρία και 3,7 στα 10 η Ρουμανία. Είναι σαφέστατο και αυτές οι χώρες θα μπουν στο Σέγγεν. Και βέβαια όχι και μάλιστα ποτέ. Πρόεδρε, τα γεγονότα δεν ψεύδονται τον Ιανουάριο έπιασαν δεκάδες τελωνιακούς στη Βουλγαρία ε, για ε, διαφθορά και λίγο αργότερα 200 Ρουμάνους τελωνιακούς. Τι θα γίνει και γίνεται και δουλεμπόριο και μόνο ε, στη Ολλανδία είχαμε πάρα πολλά κρούσματα πέρσι και να πούν στο Σέγγεν αυτές οι χώρες θα είναι έσχος και τελείως ανεύθυνο. Μπορεί να θέλουμε ό,τι θέλουμε, Πρόεδρε, αλλά να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Ανοίξτε τα μάτια σας. Δεν αξίζουν αυτές οι χώρε να μπουν στο Σέγγεν. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους εγγραμμένους ομιλητές. Ο κύριος ε, Κοβάτσεφ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο για την αντικειμενική και δίκαιη αξιολόγηση της Βουλγαρίας και Ρουμανίας και ευχαριστώ την Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποστήριξαν τον εισηγητή. Η διαδικασία αξιολόγησης της προσχώρησης των δύο χωρών θα πρέπει να υπόκειται στα ίδια κριτήρια που ίσχυαν στην αρχή ήδη το 2007. Είχαμε πει ότι από τη στιγμή που εκπληρωθούν τα τεχνικά κριτήρια από τι δύο χώρε θα γίνουν μέλη του Σέγγεν, του χώρου Σέγγεν από το 2011. Κάτι που ισχύει. Η αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων του Σέγγεν είναι ανεπιφύλακτη υπέρ τη εκπλήρωση των κριτηρίων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, παρά τι εσωτερικέ κομματικέ συζητήσει που γίνονται σε ορισμένα, σε ορισμένα κράτη-μέλη. Φυσικά θα πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μα σύνορα, να συνάψουμε συμφωνίε επανιστοχής με του Νότιου και ανατολικού γειτονέ και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μα προς χώρες που αντιμετωπίζουν τη μαζική εισρωή μεταναστών από τρίτε χώρε. Μερικοί φοβούνται ότι η μετανάστευση θα υπονομεύσει την κοινωνική πρόοδο στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά σχέδια εκτάκτου ανάγκη όπω στην Ιταλία και τη Μάλτα. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε όμω δύο διπλά μέτρα και σταθμά. Αν έχουμε κανόνε θα πρέπει να ισχύουν και στα παλιά και στα νέα κράτη-μέλη. Συνάδελφοι, η Ρουμανία και η Βουλγαρία υλοποίησαν ε, τι υποχρεώσει του, στήρισαν τι υποσχέσει του, κατέβαλαν τεράστιε προσπάθειε να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και είναι έτοιμες. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα ε, σύνορα της Μεσογείου με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο η Βουλγαρία και η Ρουμανία προστατεύουν ε, τα σύνορα της Μαύρης Θάλασσας. Το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει την απόφαση εφόσον τηρούνται τα κριτήρια ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία ήδη από φέτος θα προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν από το Σεπτέμβριο θα πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση Κοέλιο ώστε να στείλουμε ανεπιφύλακτο μήνυμα προς το Συμβούλιο ότι για να είναι ασφαλέστερα τα εξωτερικά μας σύνορα και οι πολίτες μας θα πρέπει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία να ενταχθούν από φέτος στο χώρο Σέγγεν. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι η ελευθερία των κινήσεων είναι μία από τι βασικέ ελευθερίε που απολαμβάνουν πολλοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση Και εξ ονόματο της ομάδας μου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να υποστηρίξω την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Νομίζω ότι θα πρέπει να καλωσορίζουμε τα θετικά χωρίς να ε, ξεχνούμε και να παραλείπουμε να εκφράσουμε τη λύπη μας. Ορισμένοι συνάδελφοί μας σήμερα από χώρες που έχουν προβλήματα με τη διαφθορά εκφράζουν επικρίσεις για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Μα οι δύο αυτές χώρες είναι πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να τη χάνουν ίσης μεταχείρισης. Όταν λοιπόν αύριο κληθούμε να ψηφίσουμε θα σας παρακαλούσα να ε, δείξτε την ίδια ακριβώς μεταχείριση στις δύο αυτές χώρες όπως και στη δική σας. Ευχαριστώ. Ήλτσεφ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν την Ολομέλεια πρόκειται να ολοκληρώσουμε την αξιολόγησή μας ε, για την ε, ετοιμότητα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας να ενταχθούν ε, στο χώρο του Σέγκεν. Η έκθεση του κ. Κόλλιο είναι επιτυχής και ελπίζω να τα καταφέρουμε και εμείς. Πολλοί θεωρούν ότι η αξιολόγηση του Κοινοβουλίου θα ε, ταυτίζεται με την αξιολόγηση των φιλευτέρων και σήμερα βρίσκονται εδώ οι πολίτες της ε, Βουλγαρίας και της Μανίας ε, γιατί τους έχει δοθεί το πράσινο φως και θα συνεχίσουμε ελπίζω να τους το δίνουμε. Βεβαίως δεν θέλουμε να αλλάξουν ad hoc τα κριτήρια για το χώρο του Σέγγεν. Ε, θα πρέπει να αιτιολογήσουν τη στάση τους όσοι εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί. Υπάρχουν πολλοί εδώ που ε, ήταν ε, καταρχήν σύμμαχοι των δύο χωρών και άλλαξαν γνώμη. Για ποιο λόγο ε, υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια ή υπάρχει μήπως προκατάληψη ίσως και απογοήτευση. Ελπίζω λοιπόν ότι οι Υπουργοί Δικαιοσύνη και Εσωτερικών θα συμφωνήσουν μεταξύ τους όπως συνέβη και ανάμεσα σε εμάς κατά διάρκεια της για την έκθεση Κοέλιου. Κύριε Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι στις τελευταίες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο και πιο συχνά σκεφτόμαστε με υπό τη σκοπιά των, της άμυνας των εξωτερικών σύνορων. Μερικές φορές ξεχνούμε τα εσωτερικά σύνορα. Δεν υπάρχει καμία αντικειμενική αιτία για να αντισταθούμε στην προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στο χώρο Σέγγεν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ελευθερία διακίνησης ε, των Ευρωπαίων πολιτών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημερινή συζήτηση δείχνει πόσο διχασμένη είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτοί που εγείρουν ε, ε, τεχνητά επιχειρήματα εις βάρος της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας θα πρέπει να έχουν στη συνείδησή τους και να αναλάβουν την ευθύνη της καταστροφής του ευρωπαϊκού σχεδίου. Δεν θα πρέπει να αποφύγουν μια τέτοια ευθύνη σε περίπτωση που αναχαιτήσουν αυτή την πρόσβαση. Κύριος Μπάτεν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ο χώρος του Σέγγεν ε, κινδυνεύει αυτή τη στιγμή και υπάρχουν μάλιστα και σχέδια να επεκταθεί <clears throat> στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 900.000 Ατύγκαν υπάρχουν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και πάρα πολλοί εξ αυτών θα ήθελαν να μεταναστεύσουν. Από τη στιγμή που θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στο χώρο του Σέγγεν, πολλοί εξ αυτών αναπόφευκτα θα φτάσουν στη Μεγάλη Βρετανία για να επωφεληθούν από ε, τα γενναιόδωρα επιδόματά μα ε, και το σύστημα στέγαση. Ε, σω λοιπόν σε ορισμένου να του άρεσε να συναντηθούν με τους ακτιγκανούς όταν θα φτάσουν στο Heathrow και στο Καλέ ε, να τους δώσουν τις απαραίτητες διευθύνσεις ε, για να πάνε εκεί που είναι ε, ευπρόσδεκτοι. Οι Ρωμά ίσως αλλάξουν βέβαια γνώμη για το κατά πόσο πραγματικά τελικά υπάρχουν πλεονεκτήματα στο να βρίσκεται κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Κύριος Κράης, φοβάμαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δείχνει πόσο μακριά είναι από την πραγματικότητα εάν εγκρίνει την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ε, χώρο Σέγγεν. Διαπιστώνω ότι διάφορα κράτη-μέλη ε, θα αντιταχθούν και έχουν και τους λόγους τους, πολύ καλούς λόγους. Εσύ, πρόσφατα μας λέει η Ευρωπόλ για το οργανωμένο έγκλημα σε μια έκθεσή της ότι έχουμε εγκληματικές ομάδες από την ε, Τουρκία, την Αλβανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση που θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία της εισόδου Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο Σέγγεν. Επίσης, η έκθεση αυτή ε, αναφέρεται και στην άρση υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίων για τις χώρες των Βαλκανίων. Επίσης, επιπόλαια απόφαση. Λαθρομετανάστευση από την Τουρκία θα μας έρθει μαζικά όταν μπει η Βουλγαρία στο Σέγγεν Ποιε εγγύησει μα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με τρόπο αποτελεσματικό, καμία. Τι μέτρα έχετε προβλέψει για να προλάβουμε τα περισσότερα ε, και νέα προβλήματα με Αθηγάνους και Ρωμά ε, που είναι και εγκληματικά στοιχεία πολλές φορές και πάλι καμία απάντηση. Και πού είναι τα μέτρα κατά ε, στολής και πάταξης διαφθοράς. είμαι ε, πεπισμένος ότι θα καταλάβουν και οι καλόπιστοι ότι ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε όλους τους άλλους Ευρωπαίους από το οργανωμένο έγκλημα και μαζική λάθρο μετανάστευση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαρινέσκου για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ένταξη της Ρουμανίας στον χώρο του Σέγγεν είναι ένα σχέδιο και ένα εγχείρημα που χρειάστηκε τεράστιες προσπάθειες και ανθρώπινες και οικονομικές και ε, διοικητικέ. Ε, πάνω από ένα δισεκατομμύριο έχει επενδύσει η Ρουμανία στο εγχείρημα αυτό και είναι θετικές οι ε, εκθέσεις αξιολόγησης. Έχουμε ε, πλέον ε, όλα τα κριτήρια, το εξωτερικά μας ε, σύνορα είναι από τα πιο μακρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε το πιο σύγχρονο σύστημα ελέγχου των σύνορων. Επίσης εντείναμε τη συνεργασία μας με τη Frontex. Οι επιχειρήσεις της Frontex που γίνονται στην Ελλάδα υποστηρίζονται από τη Ρουμανία. Είμαστε ο παριθμόν 2 ε, μετά τη Γερμανία ε, πάροχος και εξοπλισμού και ανθρωπίνου δυναμικού. Επίσης ε, και χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία συνεργαζόμαστε για το άσυλο και τη μετανάστευση. Η καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων και του δουλεμπορίου παρακολουθείται με βάση ε, τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Είναι μοναδική στην Ευρώπη ε, και η αντιμετώπιση του ΣΥΣ 1 και του ΣΥΣ 2. Παρακολουθούμε και τα θαλάσσια σύνορα και είναι υποδειγματική αυτή η βέλτιστη πρακτική. Και επίσης ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η Ρουμανία είναι σε θέση θεσμικά, αλλά έχει και την πολιτική βούληση για να φτάσει στους στόχους και στη δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι η ένταξή μας στο Σέγγεν δεν είναι δώρο που προσφέρεται στη Ρουμανία. Απλή αναγνώριση είναι των προσπαθειών και τον κόπο της και θα συνεισφέρει ε, προφανέστατα στην ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοέγιο και συγχαρητήρια για την έκθεσή σας. Κυρία Φαχιόν, για ένα Ευχαριστώ. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τα πολιτικά επιχειρήματα ε, να αναβάλουν ακόμα περισσότερο την ένταξη αυτή. Αυτή η εξτρεμιστική ακραία ρητορική ε, που ακούμε από τους ακροδεξιούς στο όνομα της ξενοφοβίας που θέλει να κλείσει τις πύλες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Θα πρέπει να αντιταχθούμε στην εξέλιξη αυτή και ε, να βοηθήσουμε για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Είναι απαράδεκτο τα κράτη-μέλη να θέλουν να ορθώσουν εσωτερικά σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών είναι από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης. Η διεύρυνση δε του χώρου Σέγγεν μπορεί να βοηθήσει θετικά όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποδείξουμε ότι αυτή η ιδέα της ολοκλήρωσης και της ενοποίησης είναι πολύ ζωντανή και ότι η Ευρώπη προχωρεί και δίνει το παράδειγμα και ευκαιρίες στους πολίτες. Κύριε Πρόεδρε, ε, μπορεί να άλλαξα θέση αυτήν την εβδομάδα στην ομάδα των συντηρητικών ε, και των μεταρρυθμιστών, αλλά δεν άλλαξα θέση όσον αφορά το Σέγγεν και τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Αυτό είναι το θέμα του Σέγγεν. Το θέμα είναι ότι θα αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Και η Ελβετία που είναι στο Σέγγεν, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να κλείσουν ε, τα σύνορα οι Γάλλοι δείχνει ότι υπάρχει κρίση η ε, ο ρεαλισμός δείχνει επίσης ότι θα υπάρξουν προβλήματα αν μπουν η Ρουμανία και η Βουλγαρία ε, στο χώρο του Σέγγεν. Θα υπάρχουν ε, ε, διαρροές, θα υπάρχουν κενά. Πολλοί μετανάστες θα μπορούν να φτάσουν στο καλέ χωρίς κανένα εμπόδιο. Η Βουλγαρία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Έτσι λοιπόν η πρόταση αυτή απλά θεωρώ ότι είναι πολύ βεβαιασμένη και υπερβολική. Ενώ η Ευρώπη κάνει δεν τρέχει τίποτα, ε, η έκθεση της Europol για το οργανωμένο έγκλημα το 2011 δείχνει ότι αν μπουν η Ρουμανία και η Βουλγαρία στο Σέγγεν, οι εγκληματικές οργανώσεις Τουρκίας και Αλβανίας θα επεκτείνουν τις δραστηριότητε τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ήθελα να παρθέσω λοιπόν το εξή. Η παράνομη μετανάστευση από την Τουρκία θα επεκταθεί ε, και μέσω της Βουλγαρίας. Ε, θα υπάρχει μεγαλύτερη διακίνηση των ναρκωτικών και όσον αφορά την παράνομη διακίνηση ανθρώπων αν μπουν οι δύο χώρες αυτές τότε ε, θα ε, αποκτήσουν οι Βούλγαροι και οι Ρωμά νέες ευκαιρίες ε, για ε, να προάγουν τις δραστηριότητές τους. Τέλος παρά, Στη τελική ανάλυση θα υπάρξει αύξηση της επάνω μετανάστευσης από την Τουρκία και θα υπάρχει λιγότερη ασφάλεια για τους Ευρωπαίους. Η Ευρώπη θα κάνει τη χάρη του οργανωμένου εγκλήματος. Η Λέγκα του Βορρά για μας, εμείς είμαστε αντίθετοι και αύριο όσοι υπερψηφίσουν θα φέρουν την ευθύνη μια ψήφου η οποία θα ανοίξει στο οργανωμένο έγκλημα, μια οτοστράντα, έναν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο που ε, θα ε, φέρει αυτοκίνητα που θα καταστρέψουν την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί με την αυριανή έγκριση της έκθεσης Κοέλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει ένα σαφές μήνυμα ότι αναγνωρίζει την ετοιμότητα της Ρουμανίας και Βουλγαρίας να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν. Νομίζω ότι οι χώρες αυτές έχουν ε, υλοποιήσει σημαντικά επιτεύγματα προκειμένου να ενταχθούν στο χώρο αυτό και είναι πολύ σημαντικό και για ιστορικούς λόγους, για χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης να ε, απολαύσουν αυτή τη δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα πρέπει να πληρούν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ένταξης αντίστοιχους με αυτούς που είχαν τηρηθεί από τις προηγούμενες χώρες που εντάχθηκαν στο Σέγγεν. Δεν μπορούμε να είμαστε πιο απαιτητικοί απέναντι στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία σε σχέση με τις χώρες που παλιότερα εντάχθηκαν στο χώρο Σέγγεν. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε διπλά μέτρα και σταθμά, γιατί κάτι τέτοιο υπονομεύει την ίδια τη βάση του κεκτημένου Σέγγεν, δηλαδή την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μελών. Και τα συμβάντα των τελευταίων μηνών δείχνουν ακριβώς πόσο επιτακτική ανάγκη είναι να προφυλάξουμε και να, προ... υπεραμεινθούμε των επιτευχμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεκτημένου Σέγγεν. Δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε την προσχώρηση αυτών των δύο χωρών και την αναθεώρηση του μηχανισμού Σέγγεν. Και δεν θα πρέπει οποιαδήποτε αναθεώρηση να συνδυαστεί με την ένταξη των δύο αυτών χωρών στο χώρο Σέγγεν. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον εισηγητή τον κύριο Κουέλιο γιατί ήταν πολύ επικοδομητικό το έργο του στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα όμως ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και την Ουγγρική Προεδρία για τη δέσμευσή της και την προσπάθεια που έκανε για να ενταχθούν και οι δύο αυτές χώρες στο χώρο Σέγγεν. Ευχαριστώ. Αύριο θα ψηφίσουμε για την προσχώρηση της ε, Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Νομίζω ότι είναι προφανές για κάθε δημοκράτη ότι όλες οι χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους Σέγγεν να ενταχθούν ε, σε αυτό το χώρο. Βέβαια, δεν θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί απέναντι σε ορισμένε χώρε. Θα πρέπει να ισχύουν τα διακριτήρια για όλου. Οποιαδήποτε άνηση μεταχείριση υπακούει σε πολιτικού λόγου από τη στιγμή που εξακριβώσουμε την τήρηση των ε, προϋποθέσεων από τις χώρες αυτές θα πρέπει να επιτρέψουμε την ένταξή τους ε, στο Σέγγεν. Άλλωστε ακόμη και το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά μπορεί πιο αποτελεσματικά να παταχθεί εντός του χώρου Σέγγεν υπευλήθη ένα πακέτο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να το επεξεργόμαστε γιατί το θέμα αυτό είναι κοινή πληγή ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά μόνο χαρακτηριστικά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Δεν χρειαζόμαστε κλειστές πόρτες για να πατάξουμε τέτοια φαινόμενα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ε, το αναμφίσβητα είναι κληρονομιά πολιτισμού και σήμερα λοιπόν ε, χαιρετίζουμε ένα πολύ σημαντικό πόρισμα το οποίο λαμβάνει υπόψη του τους πολίτες ε, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το σημαντικό εργαλείο. Αναφέρομαι στους πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ο χώρος του Σέγκεν θα σταθεροποιηθεί περαιτέρω και θα ενισχυθεί. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένα απτά στοιχεία πολιτισμού στην Ευρώπη και είναι ακριβώς αυτό που σας ανέφερα ότι οι Ευρωπαίοι εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια στο χώρο του Σέγγεν. Το Σέγγεν λοιπόν είναι καθοριστική σημασία για την αγορά και είμαι πεπισμένος ότι στις 24 ε, Ιουνίου αυτού του έτους ε, το Συμβούλιο ε, θα, λάβει, θα εξάγει σημαντικά συμπεράσματα θα δείξει ότι είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη. Βεβαίως θα πρέπει πριν να υπάρξει και όλη αυτή η διαδικασία της ε, ψηφοφορίας, ε, κάτι το οποίο ανέφερε και η κυρία Μάλστορμ τις τελευταίες ημέρες. Ε, η διαχείριση του χώρου του Σέγκεν σίγουρα χρήζει μεγαλύτερη συνεργασία, ενίσχυσης αλλά και επικαιροποίησης. Διαφάνεια και διάλογος, αναμφίβολα, τα κριτήρια τα έχουν καλύψει η Βουλγαρία και η Ρουμανία και συγχαίρω την, τον εισηγητή ο οποίος παρουσίασε αυτό το το έγγραφο το οποίο ε, συμμερίζονται πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, τα σύνορα της Βουλγαρίας ε, που είναι 1300 χιλιόμετρα χαρακτηρίστηκαν ασφαλή από το Σέγγεν και ε, πολλαπλές διαδοχικές κυβερνήσεις της Βουλγαρίας εργάστηκαν προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, που συνεργάστηκαν ε, σε αυτή την υπόθεση ε, για την επικοδομητική τους και ωφέλιμη στάση. Τώρα φαίνεται ότι κάποιες χώρες έχουν εφεύρει νέα εμπόδια και μάλιστα προφάσεις για την ασφάλεια και υποτιθέμενη διαφορά ε, αυτό είναι ένα θέμα. Το θέμα της διαφθοράς είναι ε, εσωτερικό της χώρας. Γι' αυτό ζητήθηκε και η παρέτηση του Υπουργού Εσωτερικών. Υπάρχει μηχανισμό συνεργασία και επαλήθευση για όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επίστροπο κυρία Μάλμστρομ για το πακέτο τη δέσμη μέτρων που πρότεινε χτε για τη διαφθορά. Η ε, Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν πρέπει να πληρώσουν τα σπασμένα των άλλων των προβλημάτων τη ασφάλεια στα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει ξενοφοβία, ο λαϊκισμό, η απογοήτευση, η αγανάκτηση να επικρατήσουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφό μου Κάρλος Κορέγιο γιατί έκανε πραγματικά πάρα πολύ σχολαστική δουλειά και ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία κάνουν σημαντικέ προσπάθειε για να ενισχύσουν τον έλεγχο των συνόρων του και το έχουν καταφέρει. Είτε πρόκειται για την αστυνομική και τη δικαστική συνεργασία για την προστασία δεδομένων, για την πολιτική θεωρήσεων και για τον έλεγχο των συνόρων κατά ξηρά θάλασσα ή αέρα. Οι τελευταίες εκτιμήσεις είναι σαφέστατες, πληρούν όλα τα τεχνικά κριτήρια. Δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε αυτή η αερα οι τελευταιε εκτιμησει ειναι σαφεστατε πληρουν ολα τα τεχνικα κριτηρια δεν μπορουμε παρα να διαπιστωσουμε αυτη Η Ρουμανία και η Βουλγαρία πλέον μπορούν να εφαρμόσουν εφαρμόσουν το κεκτημένο του Σέγγεν από πλευρά και τεχνική και ανθρώπινη στενέχωση. Ε, κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που να διευρύνει σήμερα ε, που να τη διεύρυνση του Σέγγεν. Έχουν γίνει κάποιες συστάσεις, ελπίζω να ε, τι τηρήσουν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα χερσαία σύνορα Βουλγαρία, Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί ξέρετε ότι ε, είναι αμοιβέ υποχρεώσει και πρέπει να τηρούνται. Εάν ε, μια πλευρά δεν τηρεί τις υποχρεώσεις, χωλαίνει όλο το σύστημα. Ελπίζω πάρα πολύ να συμφωνήσει το Συμβούλιο για να ενταχθούν οι χώρες αυτές στον κύκλο των προνομιούχων που είναι το Σέγγεν. Συμφωνούμε όλοι ότι έχει και μεγάλε επιπτώσει αυτό στην κοινή γνώμη και πάλι συγχαρητήρια κύριε Κοέγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. κυρία Ντανσίλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι τα κράτη που εξέφραξαν επιφυλάξεις για την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στο Σέγγεν δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι η διαδικασία αυτή είναι νομική υποχρέωση που προβλέπει η συνθήκη ένταξης των δύο αυτών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλες οι χώρες ε, υπέγραψαν τη συνθήκη ένταξης και ανέλαβαν υποχρεώσεις. Θα πρέπει ταυτόχρονα ε, όμως ε, να καταλάβουν όλες οι χώρες στην Ευρώπη ότι είναι προς όφελός τους να μπουν στο Σέγγεν η Ρουμανία και η Βουλγαρία γιατί θα συνεισφέρουμε τη σειρά τους στην ασφάλεια όλων των κρατών μελών. Η διεύρυνση του χώρου Σέγγεν είναι θετική. Θα εδραιώσει τον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. οι αποστολές τη ευρωπαϊκή Ένωση για την εξακρίβωση δηλώνουν ότι είναι καλή η σύνδεση με το σύστημα του ηλεκτρονικού Σέγγεν και ε, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ε, στο μεγαλύτερο επίπεδο. Όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν πρόσβαση ε, στα στοιχεία από την πληροφορική σε σχέση με εκείνους που θέλουν να ενταχθούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτη. Ευχαριστώ. Herr zwei Minuten. Danke, Herr Präsident. Ευχαριστώ Πρόεδρε, <clears throat> κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα Συμβουλίου. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι δύο χώρες, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, έχουν επενδύσει πάρα πολλά ε, στην διασφάλιση των νέων εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπληρούν τα κριτήρια του Σέγγεν. Οι αντικειμενικέ έρευνε που έλαβαν χώρα μέχρι τώρα κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα ότι πράγματι πληρούνται οι προποθέσει ε, για να ενταχθούν οι χώρε αυτέ στο χώρο του Σέγκεν. Ο εισηγητής μας και ο ίδιος ε, έκανε μια σχετική έρευνα επιτόπου, ήταν αντικειμενικός στην αξιολόγησή του και κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα. Κατόπιν τούτου θα συμφωνήσουμε όχι μόνο με την έκθεση αλλά και με το ότι οι δύο χώρες αυτές πρέπει να ενταχθούν στο χώρο του Σέγγεν. Ο χώρος του Σέγγεν είναι χώρος εμπιστοσύνης. Δηλαδή δεν είναι άπαξ και τελειώσαμε πρέπει να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια πρέπει να είναι διαρκείας και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες όχι μόνο για αυτές τις δύο ελπίζω λοιπόν ότι η εμπιστοσύνη αυτή θα διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα έτσι ώστε να είναι δυνατόν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ελεύθερη μετακίνηση να μπορούμε να τα διατηρήσουμε ως ένα βασικό αγαθό ε, εκείνο που με ανησυχεί βέβαια είναι μια πληροφορία που δεν μπόρεσα να επαληθεύσω. Ε, ενημερώθηκα σήμερα για αυτή την πληροφορία σύμφωνα με την οποία η Ρουμανία περιέκοψε τους μισθούς των αστυνομικών κατά ένα τρίτο. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ότι για να ε, μην δορδοκούνται ε, οι αστυνομικοί, για να εργάζονται αποτελεσματικά, ε, πρέπει να μοιβώνται και σωστά. Ελπίζω λοιπόν αυτή η πληροφορία που έφτασε σε μένα να είναι λανθασμένη και θέλω να πιστεύω ότι οι αστυνομικοί θα εξακολουθούν να υπηρετούν τη χώρα τους αλλά και την ασφάλεια του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να συνεχίσουν να αμείβονται ικανοποιητικά έτσι ώστε να μην είναι ευάλωτοι απέναντι σε κρούσματα δωροδοκίας. Ε, Επίτροπε, σύμφωνα με την έκθεση Κοέλο, η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι βάσει των αξιολογήσεων των εμπειρογνωμόνων επαρκώ προετοιμασμένε για να εφαρμόσουν τι διατάξει του κεκτημένου σέγγεν στη χερσαία θαλάσσια και εναέρια σύνορά του. τηρούν τι βασικέ προποθέσει και τα ίδια κριτήρια με άλλα κράτη μέλη για πλήρη ένταξη στον χώρο σέγγεν. στηρίζοντα την πλήρη ένταξη των χωρών αυτών επιδεικνύουμε την κοινοτική μα αλληλεγγύη και στηρίζουμε την ευρωπαϊκή ιδέα και το θεμελιώδε δικαίωμα ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών εντός της ευρωπαϊκής ένωσης δημιουργώντας μια ισχυρότερη ευρώπη όσον αφορά του προβληματισμού που τίθενται στην έκθεση για τι αυξανόμενε μεταναστευτικέ πιέσει στην ευαίσθητη περιοχή βουλγαρία τουρκία και ελλάδα αυτοί αποτελούν σύγχρονε προκλήσει για την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση και τα κράτη μέλη για να εξεύρουν ολιστικέ πανευρωπαϊκέ προσεγγίσει ώστε να ενισχύσουν αποτελεσματικά τα εξωτερικά του σύνορα να ενισχύσουν τη frontex να επιδείξουν τη δέουσα κοινοτική αλληλεγγύη και να στηρίξουν τα κράτη μέλη τη νότια ευρώπη που δέχονται τι παρανάλογε μεταναστευτικέ ροέ. ο επίκαιρο διάλογο για εξυγχρονισμό τη συνθήκη σέγγεν πρέπει να λάβει υπόψη τι πιο πάνω προκλήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, η συμμετοχή στο χώρο του Σέγγεν σημαίνει ανάληψη ευθυνών. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα πρέπει να ενταχθούν για να λάβουν τις ευθύνες τους επιτέλους. Μαζί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη για την προστασία των κοινών μας εξωτερικών συνόρων. Βεβαίως είναι το θέμα λεπτό και ευαίσθητο. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις όμως για το θέμα αυτό και σε ό,τι αφορά ε, τις ροές μεταναστών, οι ροές από τη Βόρεια Αφρική δεν διευκόλυναν τις συζητήσεις αυτές. Ωστόσο τα προβλήματα αυτά δεν θα λυθούν αν μείνουν εκτός Σέγγεν η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Το αντίθετο. Θα πρέπει ενισχυθεί η αλληλεγγύη και στην πολιτική μετανάστευση και χρειάζεται να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη σε αυτή την προσπάθεια. Όχι μόνο να μπουν λοιπόν αυτές οι χώρες, να τους επιτρέψουμε αλλά να τους επιβάλλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η Επίτροπος Μάρστρομ αναφέρθηκε στην πίστη και την εμπιστοσύνη. Βεβαίως, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να το αποδείξουν ότι μπορούν. Thank you, Chair. Το κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από ένα μήνα ήρθα δικός στις Βρυξέλλες. Στα Ουγγρικά σύνορα είδα μια τεράστια τέλειωτη σειρά 87 φορτηγών από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Δανία, την Ουγγαρία, και ήταν ε, ανταλίκε φορτωμένες με εμπορεύματα που περιμένουν οι πολίτες. Και μάλιστα καθυστέρησαν όλα αυτά τα φορτηγά από μια διαδικασία που δεν ισχύει πια στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει η προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας σε αυτό το σημαντικό χώρο Σέγγεν. Είναι σημαντικό και προς όφελος και το συμφέρον ολόκληρης Ευρώπης. Θα πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα θεσμικά της όργανα. Είπατε κύριε Επίτροπε ότι ο χώρος Σέγγεν είναι ένα σημαντικό δώρο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι και σημαντικό εργαλείο όμως για περισσότερη και όχι για λιγότερη Ευρώπη. Ε, πιστεύω ακράδαντα ότι αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υπερψηφίσει την έκθεση Κοέλιο και ελπίζω το συντομότερο δυνατό να ενεργήσει ανάλογα και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Okay, dear colleagues, I have 16. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω 16 αιτήματα τώρα για το λόγο στη διαδικασία KGI. Κατ' εξαίρεση θα σας δώσω το λόγο σε όλους, αλλά θα επιμείνω στο λεπτό. Ζητώ συγγνώμη, μόλις περνάει το λεπτό σας θα σας βίνω το μικρόφωνο. Για να μπορέσουμε να τελειώσουμε γέρο αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση Κοέγιο λέγει ότι και η Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους πλέον στο χώρο του Σέγγεν. Είναι έτοιμες οι χώρες να μπουν. Έκαναν ό,τι έπρεπε, αλλά Τώρα δεν είναι σίγουρο ε, πότε θα μπουν, διότι υπάρχουν κάποιες χώρες που διαφωνούν με την ένταξη ε, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στο Σέγγεν και τη ε, βρίσκουν προβληματική. Θα... Ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή, συνάδελφοι, και τη δική σας και του Συμβουλίου, στο γεγονός ότι η απόφαση αυτή θα έχει επιπτώσει στην καθημερινή ζωή 30 εκατομμυρίων πολιτών είναι τεράστια επιτυχία η άρση των συνόρων των ελέγχων στα ιστορικά σύνορα και έχουν κάθε δικαίωμα οι πολίτες των χωρών μας να διακινούνται ελεύθερα και να έχουν όλα τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα κάνει την Ευρώπη πολύ πιο ισχυρή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποστηρίξω ανεπιφύλακτα την ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Η έκθεση Κοέλιο δείχνει ε, καθαρά και ξάστερα ότι οι δύο χώρες πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και μία τετραετία. Φαίνεται δεν το αντιλήφθηκαν όλοι οι συνάδελφοι, γιατί ορισμένα ρατσιστικά σχόλια ε, Ευρωπαίων πολιτών εις βάρος αυτών των δύο χωρών με ανησυχούν. Δεν είμαι βέβαια τι φοβούνται ακριβώς ορισμένοι πολίτες. Πώς έχουμε πρόβλημα μετανάστευση όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται από τη μία στην άλλη χώρα της Ένωσης. Υπάρχει μία βασική και θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ισότητα. Αν υπονομεύσουμε την ισότητα θα υπονομεύσουμε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένταξή της στο χώρο του Σάνκεν είναι το επόμενο βήμα. Μετά τη Βουλγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσπαθούν προσπάθησαν να εκπληρώσουν τα κριτήρια ε, και καθυστέρησαν βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι ίδιες για όλους. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να ισχύουν και για τις δύο αυτές χώρες, ε, όπως ακριβώς και για όλες τις υπόλοιπες. Οτιδήποτε άλλο ε, θα σημαίνει διακριτική μεταχείριση. Πολλά κράτη-μέλη έχουν πρόβλημα με απιστία, δωροδοκία. Σαφώς και πρέπει να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα αυτά. Πολλοί πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουν ότι τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται μόνο σε αυτέ τι δύο χώρε. Υπάρχει και πρόβλημα μετανάστευση, αλλά πρέπει να βρούμε κάποια λύση χωρίς να ε, απαρνούμε τι τις δικές μας αρχές. Κύριε Πρόεδρε, μιλούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κρίση. Μέχρι στιγμής μιλούσαμε για την οικονομική κρίση. Αυτό που συμβαίνουν γύρω από την ε, ζώνη του Σέγγεν, φαίνεται ότι οι άνθρωποι απασχολούνται όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, γιατί μερικές φορές και αυτά διακυβεύονται. Τα γεγονότα στην Ιταλία, στη Γαλλία και στη Δανία γύρω από την ε, ε, για τη ζώνη Σέγγεν είναι ανησυχητικά. Θα πρέπει να στείλουμε ένα επιφύλακτο μήνυμα ότι δεν απειλείται η ζώνη Σέγγεν. Δεν θέλουμε τον περιορισμό τη, θέλουμε την ενίσχυση τη ζώνη Σέγγεν και τη διεύρυνσή τη. Θέλουμε ανοιχτή και όχι κλειστή Ευρώπη. Θα μα βοηθήσει κάτι τέτοιο να υπερκεράσουμε την κρίση. Και χαίρομαι που η ε, Επίτροπο έστειλε ε, ανακοινωθέν αμέσω για την κοινή μεταναστευτική πολιτική και την πολιτική ασύλου. Αλλά χρειαζόμαστε ένα επιπλέον βήμα. Θέλουμε απλώ να υπερψηφίσουμε την, την προσχώρηση Ρουμανίας και Βουλγαρίας στην ζώνη Σέγγεν, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Το. Σήμερα η Συμφωνία Σέγγεν υφίσταται μεγάλες πιέσεις από τη μια έχουμε μεταναστευτικά ρεύματα από τη Βόρεια Αφρική όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τον εκδημοκρατισμό. Ορισμένες χώρες ζήτησαν άρση προσωρινή του Σέγγεν. Άλλες χώρες για λόγους δικούς τους που δείχνουν τα στενά τους συμφέροντα ε, αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν είναι ακόμα μέλη του Σέγγεν για να τους κρατάνε ακόμα απ' έξω. Αποτέλεσμα, οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ε, βάρος των δύο παικτών. Υποστηρίζω τα θετικά συμπεράσματα της έκθεσης και επενώ για αυτά τον εισηγητή, ωστόσο δεν μπορώ να καταλάβω τους πολιτικούς λόγους για τροποποίηση των συστάσεων, γιατί στο κάτω-κάτω βάση της πολιτικής είναι ο συμβιβασμός. Δεν μπορώ να παραγνωρίσω τη νέα κατάσταση που ε, αυτά που προτείνονται ε, μπορεί να έχουν υποκειμενική ερμηνεία και προσεύχομαι στο Θεό να είμαι λάθος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι αξιολογήσεις έχουν δείξει την ετοιμότητα των δύο χωρών για την ένταξη στη ζώνη Σέγγεν και τα έγγραφα αξιολόγηση και η έκθεση δείχνουν ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπορούν να γίνουν υπόδειγμα βέλτιστων πρακτικών ε, υπό ορισμένε πτυχέ. Είμαι πεπισμένο ότι η ένταξη των δύο χωρών στη ζώνη Σέγγεν δεν θα αποβεί βάρο τη ασφάλεια των σύνορων. Αντίθετα, θα ενισχύσει την ασφάλεια των εξωτερικών σύνορων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούμε για εμπιστοσύνη. Πώ είναι δυνατόν όμω να μιλούμε για εμπιστοσύνη όταν σε ορισμένε χώρε αλλάζουν οι κανόνε του παιχνιδιού. Ορισμένε χώρε ε, ενισχύουν ε, τους κανόνες και κάνουν πιο αυστηρές τις προϋποθέσεις για την ένταξη στη ζώνη Σέγγεν. Τα επιπλέον κριτήρια που απαιτούνται από τη Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν είχαν ε, εφαρμοστεί καμία προηγούμενη χώρα. Θέλουμε ισότιμη μεταχείριση των δύο χωρών και αντικειμενική αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια. Νομίζω ότι το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι απερίφραστος προς αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, ο οποίος εκπώνησε μια έκθεση πάρα πολύ σημαντική όσο και δύσκολη γιατί είναι αντιφατικές οι θέσεις από ε, αυτού του θέματος τη ένταξη δηλαδή της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο του Σέγγεν. Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να ευχαριστήσω όλους εκείνους που κατάλαβαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται με βάση αξίες και αρχές. Η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο του Σέγγεν είναι τμήμα αυτής της ευθύνης που αναλαμβάνουν οι δύο χώρες και ανέλαβαν με την ένταξή τους το 2004 ότι θα φροντίσουν να εκπληρώσουν κάποια ε, θέματα για τα οποία είχαν δεσμευτεί και υπάρχουν εκθέσεις που το τεκμηριώνουν αυτό. Σήμερα συζητούσα με κάποιο συνάδελφο από χώρα ε, που έχει αντιρρήσεις και τον ρώτησα «Μα γιατί αντιτίθεται η χώρα» φαίνεται ότι πληρείται λέει τα κριτήρια αλλά στο εσωτερικό της χώρας ε, έχουμε λόγους εσωτερικής πολιτικής. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θεωρώ ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται στην ενιαία εφαρμογή των κανόνων. Θεωρώ ε, ε, προφανώς ότι η είσοδος της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στη συνθήκη του Σέγγεν πρέπει να είναι αποδεικτή με την τήρηση των ιδίων κανόνων που ετηρήθησαν για την εισαγωγή και άλλων κρατών στη συνθήκη αυτή. από πλευρά μου χαιρετίζω την έκθεση του συγητή του κ. Κοέλιου και την πρότασή του για την ανάγκη λήψη προσθέτων μέτρων από τη βουλγαρία για να προωθηθεί ένα ειδικό σχέδιο δράση με την ελλάδα και την τουρκία λόγω του προβλήματο τη παράνομη μετανάστευση στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. επαναλαμβάνω κύριε πρόεδρε την πάγια θέση μου ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η συνθήκη δουβλίνο ii και να λειτουργήσει το υπηρεσιακό γραφείο του frontex στην ελλάδα σε μόνιμη βάση. ευχαριστώ. Äh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το σύστημα του Σέγγεν δεν έχει. Είναι πολύ καλά νέα, πολύ ευχάριστα νέα για όσους επιθυμούν να έχουν ε, την χρήση του συστήματος ε, της ε, πρόνοιας. Εάν η Ιταλία εάν δεν εφαρμοστούν τα κριτήρια υπάρχει φόβο, η Ρουμανία και η Βουλγαρία να εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους. Το να μπουν βεβαιασμένα δύο χώρες αυτές στο Σέγγεν αυτό θα ευνοήσει το οργανωμένο έγκλημα στην Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες του Καυκάσου. Ε, καταπολεμώντας ε, τα φαινόμενα του ασύλου η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλησε να παίξει πρωτοποριακό ρόλο και γι' αυτό η Κομισιόν ανήγγειλε ότι θα υπάρχουν πιο αυστηροί έλεγχοι για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Πρέπει να είναι σαφές ότι το ΣΕΝΚΕΝ αφορά τα εσωτερικά είναι μόνο όμως αν τα εξωτερικά είναι ασφαλή. Ε, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος έχει παρακολουθήσει αυτό το θέμα γνωρίζει ότι η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Σέγγεν στην Ολλανδία είναι πάρα πολύ ακαθόδες θέμα. Έχουμε και ευρωπαϊκή ευθύνη όμως. Και υπό την έννοια αυτή έχω μια ερώτηση να κάνω στην Επίτροπο. Τι γίνεται με την εφαρμογή των κριτηρίων ε, του Σέγγεν και πώς ταιριάζει στην καταπολέμηση της διαφθοράς και τι γίνεται με τα σύνορα μεταξύ της Βουλγαρίας, λέει ο μιλητής, και της Ουκρανίας. Και τι γίνεται με τους διεφθαρμένους ε, υπαλλήλου που αφήνουν λαθρομετανάστες να περάσουν. Κάτι άλλο που είπε και ο συνάδελφος Πίρκερ. Κάνουν οικονομίες τώρα από τους μισθούς των αστυνομικών στη Ρουμανία τι γίνεται με τα κριτήρια του Σέγγεν και το συζητάνε με τα συνδικάτα των αστυνομικών. Πώς έχει κατάσταση. Μολκοβα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία τα τελευταία τρία χρόνια ε, έκαναν ε, όλα τα απαραίτητα για να καταστούν μέρος ε, μέλη του Σέγγεν. Τα μέτρα για την διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζονται αυτόματα και τα δύο κράτη εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους, γι' αυτό ανήκουν στο χώρο του Σέγγεν παρά τη μετανάστευση από την Αφρική. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όσοι έκαναν τις αξιολογήσεις πήγαν πήγαν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και διαπίστωσαν ότι και οι δύο χώρε πληρούν τα κριτήρια του Σέγγεν. Εγώ πιστεύω ότι και ελπίζω τα μέλη του Κοινοβουλίου να υπερψηφίσουν την έκθεση Κοέλιο και επίσης ελπίζω ε, το Συμβούλιο να υιοθετήσει τα μέτρα που προτείνουμε. Ε, θέλω να πιστεύω ότι και οι Βούλγαροι και οι Ρωμάνοι θα νιώσουν την ίδια χαρά που ένιωσα και εγώ όταν πέσανε τα σύνορα ανάμεσα στη Σλοβακία και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έγινε το 2007. το να επεκταθεί ο χώρος του Σέγγεν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει βέβαια καταρχήν να καλύπτονται κάποια κριτήρια. Είναι όμως και θέμα εμπιστοσύνης. Η αίτηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κατατέθηκε σε μια ενδιαφέρουσα περίοδο όταν στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται ερωτήματα για το κατά πόσον είναι σκόπιμο να υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση πολιτών. Κατά το παρελθόν άνοιξαν τα σύνορα ε, μάλλον διορθώνει η μιλήτρια, εισήχθησαν ε, έλεγχοι συνόρων για περιπτώσεις όπου είχαμε ε, παγκόσμια πρωταθλήματα, τοπικά πρωταθλήματα ή και συναντήσεις κορυφής. Αυτή τη στιγμή έχουμε αστυνομικούς ελέγχους σε εσωτερικές πτήσεις. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα είναι ότι φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου καταργείται, γίνεται κατάχρηση ε, ενός φαινομένου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Чика на място при посещенията му в България и Румъния, но израз на волята на Европейски парламент да остане. си υπάρχει какви техники πρόβλημα το οποίο Ευχαριστώ τον κύριο Κοέλιο για την ισορροπημένη και αντικειμενική του έκθεση. Νομίζω ότι το μόνο που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο αντικειμενικά η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν εκπληρώσει τα τεχνικά κριτήρια για την ένταξη στο χώρο Σέγγεν. Θα πρέπει να στείλουμε ένα σημαντικό μήνυμα, καταρχήν προς το Συμβούλιο, ότι η πρόσβαση στην, στις πληροφορίες, ο επικοδομητικός διάλογος και η λήψη υπόψη της θέσης του Συμβουλίου είναι αποφασιστική σημασίας. Γιατί το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο φαίνεται να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει το μήνυμά μας να επεκταθεί και προς τους πολίτες. Διεκδικούμε ισότιμη μεταχείριση, ίσους κανόνες για ίσα αποτελέσματα και αυτό περιμένουμε και από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κοέλιο για την έκθεσή του. Παίρνω το λόγο γιατί βλέπω ότι γίνονται απόπειρε εκμετάλλευση τη κατάσταση στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία για να λύσουν ορισμένοι τα εσωτερικά του πολιτικά ζητήματα και προβλήματα. Πριν από δέκα χρόνια τους ίδιους φόβους εξέφραζαν για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Οι τότε ηγέτες όμως δεν ήταν μειωπε και δεν έπεσαν σε αυτό το λάθος. Α θυμηθούμε το γεγονός ότι θα πρέπει να είναι οι ίδιοι οι κανόνες για όλους. Αυτό όλωστε το λέει η συνθήκη. Αρχή τη αλληλεγγύη. Η Ευρώπη σήμερα είναι πολύ διαφορετική από την Ευρώπη πριν από 20 χρόνια. Εντάξει, αλλά αν υπάρξει κρίση στο χώρο του Σέγγεν, αυτό είναι θέμα άλλη συζήτηση, όχι τη παρούση. Ε, αν χρειάζεται να αλλάξουν οι κανόνε, να αλλάξουν για όλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο ε, Κοέγιο. Πάρα πολύ καλή η εκθεσή του, ισορροπημένη όσο και αντικειμενική. Ε, είναι αποτέλεσμα ε, της γενικής τάσης και θέσεις πολλών από εμά αξίζουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία να ενταχθούν στον χώρο Σέγγεν. Προφανώς δεν θα πρέπει να φορτώνουμε σε αυτές τις δύο χώρες τα προβλήματα που υπάρχουν παντού. Παντού υπάρχει διαφθορά και αντίστοιχα προβλήματα. Ε, μπορούν όμως να ξεπεραστούν ε, με κοινή προσπάθεια αλλά και των 27 κυβερνήσεων. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ε, κατηγορούμε ορισμένες μόνο χώρες. Έχουν αποδείξει η Βουλγαρία και η Ρουμανία ότι μπορούν να εργαστούν για μια ενωμένη Ευρώπη. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος για ένα λεπτό. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία απέδειξαν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και αυτό είναι πλήρως τεκμηριωμένο από τις εκθέσεις αξιολόγησης. Και οι, οι αξιωματικοί, οι αστυνομικοί που συνελήθησαν, ε, συνελήθησαν για διαφθορά ένας ε, Ολλανδός αξιωματούχος δεν θα ίσως στην ε, ε, Ολλανδία να μην είχε συλληφθεί. Σίγουρα δεν θα διεκδικήσουμε τις πρώτες θέσεις της διεθνούς διαφάνειας, αλλά έχουμε εκπληρώσει όλα τα τεχνικά κριτήρια και αν κάποιος προσπαθεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού ενώ όσο έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, αυτό είναι παράνομο με βάση την κοινωτική νομοθεσία και ούτως ή άλλως είναι άδικο και αντιστρατεύεται και την κοινή λογική. <coughs> Εξ της Επιτροπής, η κυρία Μάλστρομ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για αυτή την πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση. Πράγματι είναι απολύτως απαραίτητο να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στο Σέγγεν ενισχύοντας τις κυβερνήσεις και τους μηχανισμούς αξιολόγησης όπως πρότεινε κατ' ουσίαν η Κομισιόν πριν από τα Χριστούγεννα και πρότεινε να ε, συμπεριλάβει περισσότερους εμπειρογνώμονες ε, και το Κοινοβούλιο σε όλα τα βήματα που θα γίνουν. Ε, είναι επίση απαραίτητο να βελτιώσουμε την βοήθεια προς τα κράτη-μέλη τα οποία για οποιοδήποτε λόγο αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πρέπει να διευκρινίσουμε τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οποίες είναι δυνατόν να επανέλθουν οι συνοριακοί έλεγχοι. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, διαφθορά. Βεβαίω και υπάρχει διαφθορά στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, αλλά υπάρχει διαφθορά και σε όλα τα κράτη-μέλη. Εχθέ μόλι η Κομισιόν κατέθεσε μία πρόταση για το πώ εμεί ε, σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τον αγώνα κατά τι ε, δορδοκέ και πολλοί από εσά το επισημάνατε αυτό. Θέλω να πω ότι έγιναν τεράστιε προσπάθειε και από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία για να ε, καλύψουν τις τεχνικές προδιαγραφές ε, ε, του Σέγγεν. Γι' αυτό λοιπόν οι χώρες αυτές πρέπει να έχουν σαφή προοπτική, σαφές πλαίσιο για το τι περιμένουμε από αυτές έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να δεχτούν τις χώρες αυτές τους κόλπους τους στην οικογένεια του Σέγγεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω όλους για τα θετικά σας σχόλια. και για τους επένους σας προς τις προσπάθειες της Ουγγρικής Προεδρίας. Ήταν σημαντικό για μας να γνωρίζουμε ότι σας έχουμε παραστάτες στο πλευρό μας. Γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλει η Βουλγαρία και η Ρουμανία να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν. Και γιατί μπορούν να ενταχθούν διότι πραγματικά έκαναν τα καθήκοντά τους. Το τελευταίο πεντάμινο και τις επόμενες εβδομάδες το Συμβούλιο που την Ουγγρική Προεδρία θα συνεχίσει τις προσπάθειές του έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας τη διαδικασία αυτή και να πούμε ε, ρητά ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι έτοιμες να μπουν στο Σέγγεν ότι ε, πληρούν ακόμα και το τελευταίο τεχνικό κριτήριο. Ε, και οι δύο χώρες έχουν καταβάλει σοβαρές προσπάθειες και αξίζουν συγχαρητήρια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης άκουσα πολλά επιχειρήματα και υπέρ και κατά της ένταξης των δύο κρατών στο Σέγγεν. Όλοι ανέφεραν ως ε, λέξεις κλειδιά την αμοιβαία εμπιστοσύνη και συμφωνώ. Η Ουγγρική Προεδρία εργάζεται ακριβώς στην οικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνης. Πώς προσπαθήσαμε να εδραιώσουμε την εμπιστοσύνη αυτή. Πρώτον, αρχίσαμε ένα διαρκή διάλογο με τις δύο χώρες, με στενή παρακολούθηση και έλεγχο των προσπαθειών τους. Προσπαθήσαμε να τους ε, βοηθήσουμε όσο γινόταν με ε, αξιολόγηση και εκτίμηση των προσπαθειών αυτών. Ταυτόχρονα είχαμε μόνιμες και διαρκείς επαφές με όλες τις υπόλοιπες χώρες που διατηρούσαν επιφυλάξεις ως προς την είσοδο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον χώρο του Σέγγεν. Προσπαθούσαμε επίσης να πείσουμε και αυτές τις χώρες να έρθουν σε επαφή άμεση επαφή με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και να ε, έρθουν σε διμερή διάλογο. Δηλαδή και παρασκηνιακά υπήρξε ε, ε, μόνιμος διάλογος και με τους δύο αυτούς εταίρους μας και προσπαθούσαμε να προαγάγουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση. Αυτή αποτελεί τη βάση για κάθε πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς τις πολιτικές αυτές δεν μπορούμε να επιτύχουμε ε, μια αρμονική απόφαση στο Συμβούλιο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Βεβαίως χρειάζεται πολύς χρόνος για να χτιστεί αυτή η αμοιβή εμπιστοσύνη. Ένα εξάμεινο έχουμε μόνο εμείς. Ελπίζω να μπορέσουμε να το φέρουμε σε αίσιο πέρα, σας είπα, και να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Και να πούν ότι μάλιστα ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους αυτές οι χώρες. Έχει γίνει αυτός ο διάλογος, οι διαβουλεύσεις, σας είπα, ε, δεν θα πρέπει να αφιστούμε προσπαθειών, όχι μόνο εμείς και οι δύο αυτές χώρες, για να δείξουν ότι είναι δεσμευμένες στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είδαμε τεράστια βελτίωση να γίνεται και πολλές προσπάθειες να καταβάλλονται από τις χώρες αυτές. Ελπίζω να συνεχίσουν έτσι και στο μέλλον. Είμαι επίση πεπισμένη ότι μπορεί να βοηθήσει κάτι ακόμα. Ακόμα και αν επίσημα δεν αποτελεί κριτήριο για την ένταξη στο Σέγγεν. Και αυτό είναι η συνεργασία και ο μηχανισμός συνεργασίας και αξιολόγηση. Τον Ιούνιο θα ε, ε, δώσει αυτή την έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μιλά για την καταπολέμηση της οροδοκίας, το οργανωμένο έγκλημα και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρατε στη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα περιγράψει αυτά, αλλά δεν είναι κριτήριο, δεν είναι μέρος των όρων. Είναι κάτι όμως που βοηθάει ε, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι μια τέτοια θετική έκθεση θα βοηθήσει σε θετική πολιτική απόφαση ή θα τη διευκολύνει. Αν με ρωτάτε τώρα για το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ατμόσφαιρα, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, ένα σύνολο πάρα πολύ ε, εξωστρεφές που ανοίγει τις πύλες του προς ε, τους πολίτες που έρχονται από το εξωτερικό. Το ακούσαμε και από τους ομιλητές σήμερα. Ορισμένοι είπαν ότι θα φύγουν από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία οι Ρωμά μόλις μπει στο Σέγγεν η χώρα τους. Μα το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών είναι θεμελιώδες δικαίωμα και θεμελιώδης ελευθερία στην Ένωση. Οι Ρουμάνοι και Βούλγαροι πολίτες ήδη από τώρα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Και εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι Ρωμά και όλοι οι πολίτες απανταχού της Ένωσης. Μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς θεωρήσεις όπου θέλουν στην Ένωση. Και είμαι πολύ περήφανη γιατί κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας εγκρίθηκε στρατηγική για τους Ρωμά που σαφώς ορίζει όλες τις ευθύνες όλων των κρατών μελών. Θα πρέπει αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του. Με καλύτερη παιδεία, με καλύτερη κατάρτιση και δυνατότητες απασχόλησης των Ρωμά θα μειωθεί η εσωτερική μετανάστευση. Και μια τελευταία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Εάν θέλει κανείς να αμφισβητήσει μια θεμελιώδη ελευθερία ή να την αρνηθεί, προς τους πιο ευάλωτους πολίτες είναι πάρα πολύ αρνητικό φαινόμενο και πάρα πολύ επικίνδυνο για την Ένωση. Αναφερθήκατε στην αθεώρηση του συστήματος. Η Ουγγρική Προεδρία ευθύς εξ αρχής εξέφρασε τις απόψεις της και είπε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο θέματα ξεχωριστά. Πρώτα την αναθεώρηση και στη συνέχεια την ένταξη αυτών των δύο κρατών, να μην αναμειγνύουμε τα δύο θέματα. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία, είναι θεμελιώδης ελευθερία στην Ένωση, να πρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα μέσα μα και να βελτιώνουμε ε, την προστασία και τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων. Γι' αυτό εργαζόμαστε τον κανονισμό για το Frontex, γι' αυτό προσπαθούμε να μειώσουμε τα μεταναστευτικές πιέσεις από τη Βόρεια Αφρική με νέα πολιτική γειτονία και γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων για να αυξηθεί η χρηματοδότησή της. Είμαστε στο τελευταίο βήμα τώρα και μπορούμε, πιστεύω, να φτάσουμε σε συμφωνία. Είναι το γνωστό πρόβλημα των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων παρόδο. Λοιπόν, ας αναθεωρήσουμε το Σέγγεν, να δούμε πού χρειάζεται αναπροσαρμογή, πού χρειάζεται ρύθμιση, αλλά ε, βήμα-βήμα και με τη σειρά τα βήματα. Κυρίες και κύριοι, Είμαι πεπισμένη ότι η αναθεώρηση του χώρου του Σέγγεν και η διεύρυνσή του θα λυθεί μεθαύριο στη συνεδρίαση του Συμβουλίου και ελπίζω να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις ε, για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Ευχαριστώ. Τέλος, ο εισηγητής μας, ο κύριος Κοέλιο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, ένα συνάδελφο είπε ότι το να αφήσουμε την ε, Ρουμανία και Βουλγαρία να μπουν στο Σέγγεν θα ήταν πεθαριώδη απόφαση. Διαφωνώ ριζικά. Εμείς ε, εκτιμούμε μόνο τα λογικά επιχειρήματα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ενηλίκων, και μάλιστα τη σορθή επιχειρηματολογία και τη δίκαιη επιχειρηματολογία. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε κατά πόσο η Ρουμανία και η Βουλγαρία πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο Σέγγεν και αν εφόσον τις πληρούν θα πρέπει να ενταχθούν. Είναι ε, φυσικά λογικό και οι πολίτες τους να αναγνωρίζονται ως ισότιμοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει οι πολίτες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας να γίνουν όμοιροι πολιτικών συζητήσεων. Είμαστε υπέρ ενό νέου συστήματο αξιολόγηση του Σέγγεν, γιατί υπάρχουν μερικέ αδυναμίε στο χώρο Σέγγεν, για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, για να τα επιλύσουμε ή να είμαστε σε θέση να λάβουμε κάποιε αποφάσει εφόσον ε, παραμένουν αυτά τα προβλήματα. Οι συζητήσει όμω για το νέο σύστημα αξιολόγηση του Σέγγεν δεν μπορεί να αποτελέσει το πρόσχημα για να καταστήσουμε όμοιρους αυτής της νομοθετικής διαδικασίας τους πολίτες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Είναι διαφορετικές αυτές οι διαδικασίες, θα πρέπει καθεμία να ακολουθήσει το ρυθμό της. Ευχαριστώ την Υπουργό Γκιόρη ε, για, το σχόλιο της ε, για την Πορτογαλία και διευκολύνθηκε πραγματικά στην Προεδρία μας η η προσχώρηση της δικής σας χώρας και άλλων χωρών στη ζώνη Σέγγε. Σας ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο και την υπεθύμηση. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσει η συζήτηση και πιστεύω ότι με το αποτέλεσμα της αυριανής ψηφοφορίας θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο ότι όταν το Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί του πολίτε τη Ευρώπη με ευελπιστώ μεγάλη πλειοψηφία πει ναι στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία ελπίζω κάτι αντίστοιχο να πραγματοποιήσει το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ τον εισηγητή μας τον κύριο Κοέλιο. Νομίζω ότι μετά την συντριπτική πλειοψηφία των θετικών σχολείων που ακούσαμε σήμερα στη συζήτηση από τους Ευρωβουλευτές αλλά και από τις θετικέ αξιολογήσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής ε, θα ήθελα να συγχαρούμε θερμά την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Στις 12 το μεσημέρι. Συνάδελφοι, ένα-δύο λεπτά διάλειμμα για να περάσουμε αμέσως μετά στο, στην ώρα ερωτήσεων προς την Επιτροπή.